Buenos Ας αρχίσουμε αν θέλετε. Απέναντι στα τελεσίγραφα, τους εκβιασμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Κομισιόν και των Ευρωπαίων ηγετών και μπροστά στις απειλές αυτές ένα κύμα λεγγύης ξεπηδά για να σταθεί δίπλα στον ελληνικό λαό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρισκόμαστε σήμερα με τον σύντροφό μας Δημήτρη Παπαδημούλη, με άλλους συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ενωτική Αριστερά και άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Ευχαριστώ τον Τζόρντι Σεμπάστια και τον Τέρε Κάμπρας για την παρουσία τους εδώ. Αυτό που κατανοούμε είναι ότι διακυβεύεται η ίδια η δημοκρατία δεν τίθεται πλέον θέμα υπέρ ή κατά του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ ή κατά του Τσίπρα. Μιλούμε για αξιοπρέπεια, για δημοκρατία απέναντι σε δικτατορικές επιταγές. Εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη στηριγμένη στη βούληση των λαών και όχι στηριγμένη σε μια Ευρώπη των χρηματαγορών. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδειξαν ότι αλλά για την δημοκρατία. Δεν ενδιαφέρονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεξάγει αγώνα κατά της λιτότητας που θίγει τους φτωχότερους και πλέον ευάλωτους στην Ελλάδα. Οι Έλληνες αποφάσισαν να ξεσηκωθούν και γι' αυτό τους τιμωρούν γι' αυτό είναι θύματα ενός πραξικοπήματος. Σιωπηρού βέβαια, δεν είναι τα τάγκ στους δρόμους, πρόκειται όμως για πραξικόπημα. Γιατί θέλουν τελικά αυτοί που κάνουν το πραξικόπημα να ανατρέψουν την κυβέρνηση που εκλέχθηκε, που είναι η μόνη ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία ξεσηκώθηκε κατά της Μέρκελ, της Bundesbank, κατά των ελίτ. Γιατί αποφάσισαν το μέλλον τους, τη ζωή τους, εκείνη των μελλοντικών γενεών, να μην ε, δεχτούν να παρετηθούν από αυτές υπέρ των οικονομικών συμφερόντων. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα, να μην ξαναγίνει αυτό. Κανένας ευρωπαϊκός λαός να μην βρεθεί στην ίδια κατάσταση υπό του κεφαλαίου. Και είναι ένα μήνυμα προς το Ισπανικό κράτος. Γιατί οι επόμενες εκλογές που θα έχουμε εκεί πρέπει να σταματήσουν την κατάσταση αυτή. Τον Μάιο στην Ισπανία δώσαμε ένα μήνυμα. Ο Ραχώη πρέπει να φύγει από τη Μουκλώα. Η αλλαγή θα γίνει και γι' αυτό θέλουμε να στείλουμε το μήνυμά μας κατά όλων των εκβιασμών και όλων των πιέσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή σε βάρος του ελληνικού λαού. Αλλά και εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η Ελλάδα δεν θα είναι η μόνη φωνή αξιοπρέπειας στην Ευρώπη. Θα ακουστούν πολύ περισσότερες. Και θέλω να εκφράσω και πάλι την αλληλεγγύη μας προς τον ελληνικό λαό και με αυτό θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ στη Γκουε που μας προσκάλεσε εδώ. Είμαστε από τους πράσινους και θέλουμε και εμεί να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα προ τον ελληνικό λαό και την ελληνική κυβέρνηση που δημοκρατικά εκλέχτηκε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Βαλένθια και ήμουνα με έναν σύντροφο εκεί, ο οποίο σπουδάζει και μου είπε «Εσύ που είσαι στην Ευρώπη, για εξήγησέ μου λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν, επιστρέφουν τα, δεν επιστρέφει τα χρήματα που έχει δανειστεί». Και είπα ότι δεν είναι δικό του δαν, δεν είναι σωστό. Και εξήγησα. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι ποιο θα πήρε τα χρήματα αυτά. Σκέψου ότι είπε να είσαι σε μια τάξη, να σου έχει δανείσει κάποιο χρήματα και να τα παίρνει καραμέλες και να μην τα παίρνει για αυτό για το οποίο τα ζήτησε. Και μετά να μην. Να, πρέπει όλη η τάξη να ξεπληρώσει τα χρήματα αυτά. Εντάξει, με κάθε αναλογία. Τώρα είμαστε στην Ευρώπη και το μήνυμα βγαίνει με τέτοιο τρόπο που η κοινή γνώμη θέλουν να καταλάβει πως έχει αποτύχει ο ελληνικός λαός και ότι υπάρχει κάποιος που είναι καλός, η Τρόικα, που θέλει να του σώσει. Νομίζω ότι αυτή η αντιστροφή της πραγματικότητας πρέπει να φανεί ότι δεν είναι αλήθεια. Αυτός που έχει αποτύχει είναι η οικονομική πολιτική της Τρόικας, η οποία προσπάθησε να έχει κέρδη με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και παίρνοντας τις αποταμιεύσεις ε, των λόν του Νότου και του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν ο τρόπος ε, που βγαίνουν τα μηνύματα δεν είναι σωστή. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα μέτρα τα οποία προσπαθούν να επιβληθούν στους Έλληνες τη μείωση των συντάξεων κτλ. είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ήδη μέχρι τώρα έχουν γίνει και έχουν χειροτερέψει την κατάσταση του ελληνικού λαού. Τρόικα θέλει να βγάλει από πάνω της την ευθύνη, ενώ η Τρόικα είναι εκείνη η οποία οδήγησε σε αυτή την κοινωνική καταστροφή με την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που έχουμε καταδικάσει και καταγγείλει επανειλημμένως. Με την Μαρίνα συμφωνώ. Η περίπτωση της Ελλάδας δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αποτελεί σύμβολο της αντίστασης αυτού του τύπου της πολιτικές που είναι η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και μπορεί να αλλάξει. Εγώ είμαι αισιόδοξο και συμφωνώ μαζί της ότι οι τελευταίες εκλογές που έχουν γίνει σε επίπεδο αυτόνομης περιφέρειας αλλά και αλλού, αυτό ακριβώς δείχνουν. Η κατάσταση σήμερα δεν είναι μόνο το θέμα της επιβίωσης, επιβίωση του ελληνικού λαού, ενώ έτσι, που έχει εγκαταληφθεί και που δεν έχει καν τις βασικές υπηρεσίες στη διάθεσή του, αλλά μιλάω και για την ίδια την ιδέα της Ευρώπης. Διότι στην πραγματικότητα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να δουλεύουν υπέρ της ευημερία των ευρωπαϊκών λαών. Αν λοιπόν η Ελλάδα δεν τα καταφέρει με την αλληλεγγύη των υπολείπων να αποφύγει αυτήν την, ε, αυτό το πνίξιμο που τις κάνουν, τότε θα πληγούν και άλλοι. Από πλευρά της ε, Τρόικα έτσι εξαφανίζεται η Ευρώπη, γιατί δεν έχει νόημα αν δεν μπορεί να βοηθήσει το κόσμο. Δεν μπορεί λίγοι να κερδίζουν και όλοι οι υπόλοιποι να χάνουμε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την αλληλεγγύη μα προ τον ελληνικό λαό και την κυβέρνησή του, που έχει εκλεγεί νόμιμα. Επιμένω σε αυτό. Πρόκειται για μια δημοκρατία που ενοχλεί βέβαια κάποιου επειδή προσπαθεί να πετύχει τη συμμετοχή του κόσμου για να αποφασίσει. Επιμένω λοιπόν ότι πρόκειται εδώ πέρα για μια στρέβλωση της ιστορίας που μας έχουν πουλήσει τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ. Είμαι ο Μελούρμπαν από το παδέμος Είμαστε πολλοί εδώ, γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω απλώ να πω ότι πιστεύω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας δίνουν μαθήματα δημοκρατίας σήμερα. Γιατί η δημοκρατία είναι ερωτήσεις είναι επιλογές. πολύ; όταν είπαν στον Θαπατέρο να ολοκληρώσει το εκλογικό του πρόγραμμα και να εφαρμόσει τις χειρότερες περικοπές που έχουμε ποτέ ζήσει στην Ισπανία, αποφάσισε να δώσει σημασία στο λαό που τον ε, εξέλεξε η δημοκρατία αποφασίζει. Αυτό θα θέλαμε να έχει γίνει λοιπόν με το Θαπατέρο. Και όταν ε, το 135 το άρθρο του συντάγματος άλλαξε για να πληρώσουμε τα χρέη μας, καταρχήν, κατά προτεραιότητα, αγνώντας τα δικαιώματά μας, ε, θα θέλαμε να μας είχαν ρωτήσει αν συμφωνούμε πριν το αποφασίσουν. Μία κυβέρνηση με αξιοπρέπεια, μια κυρίαρχη κυβέρνηση ρωτάει, ρωτάει το λαό της πρώτα. Και αυτό ακριβώς είναι που ενοχλεί σήμερα. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και αλλιώς και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μας δίνουν μάθημα δημοκρατία σήμερα. Και πάλι. Και μας δίνουν και μάθημα κυριαρχίας, λαϊκής κυριαρχίας. χωρίς να επηρεάζεται η πολιτική που λέει ότι η μοναδική λύση είναι να συνεχίζουμε να πλήττουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, τα πιο βασικά ενός λαού, ο οποίος έχει τιμωρηθεί ξανά και ξανά. Από την αρχή της εφαρμογής των μέτρων, ο ελληνικός λαός έχασε το 25% του έπτου. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να υπογραμμίζουμε. Η κυριαρχία λοιπόν αυτό ακριβώς σημαίνει ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε τέτοια μέτρα τα οποία αντιβαίνουν προς τα συμφέροντα του λαού σου. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό που έγινε ήταν εκβιασμός. Και με τους εκβιασμούς ποτέ μα ποτέ δεν μπορεί κανείς να καταλήξει σε καλή συμφωνία. Άμα υπάρχουν εκβιασμοί, σπάει. Στα Ηνωμένα Έθνη, για παράδειγμα, ετοιμάζουν ένα πρωτόκολλο για την αναδιάστρωση κυρίαρχων χρεών. Και λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση χωρίς ε, σταμάτημα πληρωμών. Συμφωνία δηλαδή για πάυση πληρωμών ε, χρεών. Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, υπήρξε μια συνεχής απέτηση πληρωμών η οποία οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτό που ενδιαφέρε δεν ήταν να πληρωθεί το χρέος, αλλά να σπάσει μια κυβέρνηση η οποία είχε εκλεγεί νόμιμα, είχε βγει από την κάλπη νόμιμα. Είναι ανεύθυμος ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν και το Δουνουτού και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οδήγησαν σε 40 ε, δις ε, ευρώ απώλειες. Ενώ ήταν μόνο με ένα δις 600, 600 ε, εκατομμύρια η διαφορά. Τώρα έχει βρεθεί η κυβέρνηση ελληνική σε μια κατάσταση που λέει ότι μπορεί να υπάρχει διαφορετική λύση. Υπάρχει διαφορετική λύση και είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε για να μην δεχόμαστε μια πολιτική η οποία πνίγει τον κόσμο, η οποία καταστρέφει τα συμφέροντά μας. Εντάξει, σώζουμε τράπεζες. Όχι. Ανθρώπους πρέπει να σώζουμε, λαούς πρέπει να σώζουμε. Έχει την πλήρη αλληλεγγύη μας ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Καλημέρα και από μένα. Έχω βραχνιάσει, συγγνώμη. Είμαι ο Δικάπρας, ευρωβουλευτής από την Καταλωνία. Συμμετέχω και εγώ στην ομάδα των Πρασίνων, όπως και ο συνάδελφος που μίλησε πριν. Όλα αυτά που λέτε, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα, δεν χρειάζεται να προσθέσει κανείς σε πολλά πράγματα. Δύο σημεία θέλω να θίξω. Το ένα είναι ότι έχει μεγάλη σημασία το δημοψήφισμα ο λαός να μπορεί να αποφασίσει αυτό που θέλει. Είναι και αυτό που εδώ και τόσο καιρό λέμε στην Καταλωνία, ότι θέλουμε να μπορούμε να αποφασίζουμε μόνοι μας. Ναι, βεβαίως και οι λαοί έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν από μόνοι τους και να αποφασίζουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για τους εαυτούς τους και μάλιστα σε στιγμές τόσο δύσκολες και κρίσιμες. Όμως και κάτι ακόμα. Υπάρχει κάτι που φοβάμαι. Παρόλο που ίσως σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να συμφωνήσει γιατί τώρα βλέπει το πρόβλημα που δημιουργείται, που έχει μπροστά της, όμως φοβάμαι ότι δεν θα καταλήξουμε σε κατάλληλη και επαρκή συμφωνία, γιατί δεν θα λαμβάνει υπόψη αυτό το μνημόνιο για την μη πληρωμή του χρέους. Και επιτρέψτε μου και για κάτι ακόμα, αυτό το μορατόριο Εδώ νομίζω ότι όντως πρέπει να διαγραφεί ένα μέρος του χρέους. Γιατί η χρέωση της Ελλάδας θα συνεχιστεί για αιώνες. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα το οποίο δεν αναφέρει κανείς και μου κάνει εντύπωση. Το 1953 αυτοί που κέρδισαν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βρεθήκαν στο Λονδίνο και αποφάσισαν, πήραν την απόφαση του Λονδίνου για τη Γερμανία ακριβώς. Και εκεί υπολόγισαν το χρέος της Γερμανίας από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το χρέος της Γερμανίας από τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τα πρόσθεσαν όλα αυτά λοιπόν. Προσοχή, ε! Η Γερμανία πήρε και σχέδιο Μάρσαλ, έτσι, αλλά αυτό δεν το βάζω στην πάντα. Και είπανε λοιπόν ότι έπρεπε να πληρώσει αυτό το χρέος η Γερμανία. Αλλά αυτό που δεν λέμε ποτέ είναι ότι η Γερμανία τελικά 3 Οκτωβρίου του 2010 πλήρωσε τελικά το χρέος της η Γερμανία. 3 Οκτωβρίου του 2010 έγινε αποπληρωμή. Συνεπώ, ποια είναι τα μαθήματα που παίρνουμε. Πρώτον, ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να γίνει τέτοια αναδιάρθρωση, επιμήκυνση, ε, περικοπή, ό,τι θέλετε. Δεύτερον, στην περίπτωση της Γερμανίας, η οικονομική δύναμη της Γερμανίας καθυστέρησε τόσο πολύ, που είναι τόσο μεγάλη οικονομική δύναμη, έτσι. Η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει, γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει διαγραφή ένα μέρος σημαντικό του χρέους πρέπει να διαγραφεί. Τα υπόλοιπα θα είναι μικρά, μικρές διορθώσεις. Κατά τα άλλα όλοι μας την ελληνική προς τον ελληνικό λαό. Αυτός υποφέρει, αυτός δυσκολεύεται. Και αυτός είναι που πρέπει να αποφασίσει. Ευχαριστούμε. Δημήτρη. Ευχαριστώ Μαρίνα. Λέγομαι Δημήτρης Παπαδημούλης, είμαι Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους από ένα ευρύ φάσμα της ευρύτερης αριστεράς και των πρασίνων, των Ποδέμος, για την ε, έκφραση αλληλεγγύης τους. Είναι αλληλεγγύη όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό. Στη μάχη που δίνουμε για δημοκρατία, για αξιοπρέπεια, εναντίον της λιτότητας για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στην Ευρώπη, για μια διαφορετική Ευρώπη που να υπηρετεί τους πολίτες και όχι τις τράπεζες και τους τραπεζίτες. Οι επόμενες ώρες είναι ιστορικής σημασίας και οι ευθύνες των Ευρωπαίων ηγετών είναι τεράστιες. Δεν είναι ώρα για εκβιασμούς, δεν είναι ώρα για τελεσίγραφα, γιατί αυτά ήδη απειλούν όλη την Ευρώπη με ένα τεράστιο κόστος και τους ευρωπαϊκούς λαούς με πρόσθετο κόστος πέρα από αυτό που έχει προκαλέσει μια άγρια λιτότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι ακόμη και τώρα, ακόμη μέσα και στις επόμενες ώρες για μια βιώσιμη συμφωνία η οποία να εξασφαλίζει τον τερματισμό της λιτότητας χωρίς νέα ελλείμματα με μια αξιόπιστη συμφωνία για τα δημόσια οικονομικά αλλά και με μια σαφή δέσμευση για απομείωση του μη βιώσιμου χρέους καθώς και ένα αναπτυξιακό πακέτο που αναξιοποιεί διαθέσιμους και νέους ευρωπαϊκούς πόρους που να επιτρέψει στον ελληνικό λαό να ελπίζει, στην ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί, στην ελληνική κοινωνία να επουλώσει βήμα-βήμα τις πληγές που προκάλεσαν όλα αυτά τα χρόνια με την άγρια λιτότητα. Ένα από τα μεγάλα μας επιχειρήματα, ένα σημείο που μας δίνει δύναμη είναι η αλληλεγγύη των, ενός μεγάλου τμήματος των ευρωπαϊκών λαών και ιδιαίτερα των λαών του Νότου, του λαού της Ισπανίας, η απάντηση που θα δώσουν τις επόμενες ώρες οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον αγώνα για δημοκρατία και αξιοπρέπεια που κάνει ο ελληνικός λαός είναι ένας καθρέφτης, είναι ένα κριτήριο, είναι λιδία λίθος όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες για το πώς θα αντιμετωπίσει η ίδια η Ευρώπη τα δικά της προβλήματα. Γιατί η συνταγή της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού έχει αποτύχει παταγωδός. Χθες η διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωκοινοβουλίου ομόφωνα ζήτησε παράταση του ισχύοντος προγράμματος στην Ελλάδα και επίγουσα επανέναρξη των συνομιλιών έτσι ώστε ακόμη και σήμερα να υπάρξει αυτή η βιώσιμη λύση για την οποία εργάζεται η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει ακόμη καιρός. Ελπίζω με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της διεθνούς οι Ευρωπαίοι ηγέτες να καταλάβουν ότι δεν είναι ώρα για εκβιασμούς, είναι ώρα για δημοκρατία και για στροφή από τη λιτότητα στην ανάπτυξη. Ο αγώνας για αξιοπρέπεια που δίνει ο ελληνικός λαός, ο αγώνας για ελπίδα, έρχεται αντιμέτωπος με τα σχέδια για να μετατραπεί η κυβέρνηση Τσίπρα σε μια σύντομη αριστερή παρένθεση. Πρέπει να αποτύχει αυτό το σχέδιο, πρέπει να παραμείνει η ελπίδα ζωντανή, πρέπει να τελειώνουμε με τη λιτότητα, πρέπει να αναπτύξουμε τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Θέλω να αποφεληθώ για να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συντροφού που είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά που βρίσκονται μαζί μας και τις βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σακοράφα και την κυρία Κούνεβα αλλά και τον ε, το Στέλιο. Μέχρι τη μία έχουμε κανονικά την αίθουσα αλλά φαντάζομαι 10 λεφτά και ακόμα μπορούμε για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να, να καταλάβω καλά. Υπάρχει περιθώριο για συμφωνία πριν από αύριο και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά να τη ρωτήσουμε θα απογοητευτούν αν δεχτεί συμφωνία πριν από το δημοψήφισμα ο Τσίπρας και πώς αυτό θα επηρεάσει τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιήσετε την κατάσταση στην Ελλάδα για να δείξετε πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ. Η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή επιδιώκουν μια βιώσιμη συμφωνία που να επιτρέψει στην Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη, να αναπτυχθεί, να κάνει αυτές τις αλλαγές που χρειάζεται, αλλά για να επιτευχθεί αυτή χρειάζεται εκτός από νοικοκυρεμένα, ισορροπημένα δημόσια οικονομικά, απομείωση του χρέους και ένα αναπτυξιακό πακέτο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη ακόμη και σήμερα να αξιοποιήσει την έκκληση του Ευρωκοινοβουλίου για να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία. Και η Ευρωομάδα της Αριστεράς σύσσωμη υποστηρίζει τον αγώνα της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν θέλουμε μια συμφωνία υποταγής, θέλουμε μια βιώσιμη συμφωνία που να επιτρέψει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί αλλά και σε όλη την Ευρώπη να αλλάξει ρότα. Και στους ευρωπαϊκούς λαούς του Νότου που υποφέρουν από αυτή την άγρια μορομερή λιτότητα να υπάρξει ελπίδα. Αν το πετύχουμε αυτό δεν θα είναι αρνητικό για τις δυνάμεις της αριστεράς και των πρασίνων στην Ισπανία ή στις άλλες χώρες θα είναι μια επιβεβαίωση ότι υπάρχει αναλλακτική λύση. Νομίζω ότι αυτό που θα φανεί είναι ότι όταν μια κυβέρνηση δεν γονατίζει, δεν κατεβάζει τα χέρια και προσπαθεί να πετύχει, πετυχαίνει κάτι για τον κόσμο, για το λό. Γιατί πάντα από την Ευρώπη μας λέγανε περικοπές και κανέναν επίτροπο. Τώρα, πέρα από αυτά, όταν πραγματικά διαπραγματευόμαστε υπέρ των συμφερόντων της πλειοψηφίας, τότε βγαίνουν πράγματα από τα οποία υποφελείται η πλειοψηφία. Και ο κίνδυνος είναι και αυτούς που κερδοσκοπούν. Φυσικά πρέπει να φοβούνται αυτοί, γιατί δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να κερδοσκοπούν όπως κάνουν τώρα. Το 77% των χρημάτων έχει πάει στις τράπεζες. Ε, αυτό τελείωσε. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖ όλους αυτούς τους μήνες αυτό που δείχνει είναι ότι κυβερνάει με το μυαλό στο λαό. Και αν πετύχουν μια συμφωνία, η συμφωνία αυτή ποτέ δεν θα είναι μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε ασφυξία το λαό όπως οι συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και γι' αυτό και πολύ θα χαρούμε αν τελικά επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Και καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια συμφωνία η οποία δεν οδηγεί σε φτώχεια, σε ανεργία και σε μιζέρια τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Για την ερώτησή σας, εμείς οι δικές μας πολιτικές ε, δυνάμεις και οι πράσινοι που όλοι βρισκόμαστε εδώ για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στην Ελλάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξηγήσουμε ότι η ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάδα αυτό το οποίο δείχνουν είναι ότι με αξιοπρέπεια, με θάρρος, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους ισχυρούς με θάρρος και αξιοπρέπεια, μπορούμε να μην μένουμε γονατισμένοι μπροστά στο μεγάλο κεφάλαιο τους ισχυρούς και τις τράπεζες. Αυτό δείχνει και ο αγώνας του ελληνικού λαού, που είναι ένας αγώνας τον οποίο συμμεριζόμαστε εμείς από την αριστερά στην Ισπανία και αυτό ακριβώς είναι που θα εξηγήσουμε στον κόσμο. και εγώ παρόλο που δεν απευθυνθήκατε σε μένα, αλλά στην προεκλογική εκστρατεία πολλές φορές είπαμε στη Βαλένθια ότι αν είχαμε το δικό μας βαρουφάκι και κερδίζαμε τις εκλογές εντάξει δεν μιλάω απαραίτητα για καθηγητή οικονομολόγο αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε την αξιοπρέπεια να μην συμμετέχουμε στις πολιτικές λιτότητας μας ε, επέκριναν πολύ. Αλλά τι έγινε με τις εκλογές. Ο κόσμος δηλαδή καταλαβαίνει ότι η θέση της Ελλάδας δεν είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να οδηγήσει τη χώρα σε χάος. Κάθε άλλο. Να το αποφύγει. Παρακαλώ. Λουθαγιάννα από το Ελπαΐς. Στον κύριο Παπαδημούλη, θέλω να σα ρωτήσω, βλέπετε αυτή τη στιγμή να γίνονται διαπραγματεύσει ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη συμφωνία από όλε τι πλευρέ. και για το πακέτο ανάπτυξη που ακούσαμε χθε με την πρόταση του κύριου Γιούνκερ. Υπάρχει ένα πακέτο επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα, σωστά. Πιστεύετε ότι είναι επαρκέ. θεωρείτε ότι φτάνει ή όχι. Ευχαριστώ την ώρα που μιλάμε και μέχρι να τελειώσει το ισχύον πρόγραμμα τα μεσάνυχτα ε, της Τρίτης, σήμερα, 30 Ιουνίου, υπάρχει και χρόνος και γίνονται και προσπάθειες για να υπάρξει μία συμφωνία έτσι όπως την επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση αλλά την έχει ανάγκη και συμφέρον και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα ομόλογα στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, με την πορεία του, δημόσιου χρέους. Το κοινό συμφέρον και η κοινή λογική απαιτεί να δοθούν απαντήσεις και λύσεις που να δίνουν ελπίδα και αξιοπρέπεια στους Έλληνες πολίτες και όχι ταπείνωση. Όχι ένα μήνυμα ότι όποιος ψηφίζει διαφορετικά προς τα αριστερά πρέπει να τιμωρείτε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε κάθε λεπτό για μια τέτοια συμφωνία, ακόμα και μέσα στην ημέρα. Αυτό που δεν είμαστε διατηθειμένοι είναι να σκύψουμε, να γονατίσουμε, να υποταγούμε και να δεχθούμε την όποια συμφωνία ανεφόρων. Και για το πακέτο που ρωτήσατε, υπάρχει ανάγκη πέρα από τους διαθέσιμους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων να εξασφαλιστούν και νέοι πόροι από νέα σχήματα όπως το Ταμείο Γιούνκερ και κυρίως η εμπροστοβαριστούς αξιοποίηση για να δοθεί επιτέλους μια όθηση αναπτυξιακή στην ελληνική οικονομία που έχει καταστραφεί με μια ύφεση που υπερβαίνει το 25%. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Μετά από χρόνια η Ισπανία έχασε το ρεκόρ στην ανεργία. Το πήρε η Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Και γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. στα αγγλικά. Κύριε Παπαδημούλη, εάν ο ελληνικός λαός πει όχι την Κυριακή, θα δεχτεί τότε την ευρωπαϊκή πρόταση η κυβέρνησή σας ή θα παραιτηθεί. No. The, the answer is no to, uh, uh, sorry, yes. Ναι, ναι, καταλάβατε πάντως εάν πει ναι, ναι, εάν πει ναι στη Ναι. Πέρα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα υπάρχει ανάγκη επανέναρξης των συνεμιλιών για μια συμφωνία. Όσοι λένε ότι ναι σημαίνει ευρώ και όχι σημαίνει δραχμή, δεν λένε αλήθεια. Κρύβουν την πολιτική τους επιδίωξη που είναι να γίνει η κυβέρνηση Τσίπρα μια σύντομη αριστερή παρένθεση κρύβουν την πρόθεσή τους να τιμωρεθεί ο ελληνικός λαός γιατί ψήφισε όχι στη λιτότητα, γιατί ψήφισε μια διαφορετική κυβέρνηση. Η απάντησή μας είναι ότι εφόσον το δημοψήφισμα βγάλει ένα αποτέλεσμα, θα επηρεάσει αυτό την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Και φυσικά αν η απάντηση είναι ναι, τότε θα δυσκολευτεί η προσπάθεια της Ελλάδας και του ελληνικού λαού να, να πετύχει μια αξιοπρεπή συμφωνία. Επαναλαμβάνω όμως κάτι που είπα και πριν, εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμη και σήμερα για μια βιώσιμη συμφωνία, πριν την Κυριακή. Αρκεί και η άλλη πλευρά να δείξει το ρεαλισμό που δείχνει η κυβέρνηση Τσίπρα. Όχι, απλώς θέλω να ξέρω, οι ισπανικές ομάδες μήπως μπορείτε να μου πείτε αριστερά πώς θα αντιδράσει στις επικρίσεις που σας έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Ισπανία. Κατά κάποιο τρόπο το είπαμε. Ο Ραχόη τι μας έφερνε κάθε φορά από την Ευρώπη. Έναν επίτροπο. Και ένα πακέτο μέτρων που ήταν τελικά αρκετά καταστροφικό από ό,τι είδαμε. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Μας έφερνε ένα πακέτο μέτρο που τι έλεγε περικοπές, ε, αύξηση ΦΠΑ, στο φως, στο ψωμί, στο γάλα και αφαιρούσανε ΦΠΑ από τα γιότ. Τώρα εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει κανείς. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ένα μάθημα δημοκρατίας από πλευράς του ελληνικού λαού και από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης που αντίθετα από άλλες κυβερνήσεις οι οποίες εφάρμοζαν τόσο μεγάλες περικοπές το έκαναν χωρίς να ρωτάνε κανέναν. Έπαιρναν διακοπές και, ε, διαταγές και τελείωσε. Ενώ τώρα η κυβέρνηση ρωτάει το λαό. Δεν είναι δυνατόν όμως όταν βλέπουμε ότι ανεβαίνει η δημοκρατία να πέφτουν τα χρηματιστήρια. Ε, δεν είναι δυνατόν. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ακριβώς αυτό. Ότι ενισχύεται η δημοκρατία στην Ελλάδα και ξαναβρίσκουν, ξαναδίνουν αξιοπρέπεια στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη που βλέπουμε που κάνει τον εκβιασμό στην Ελλάδα δεν είναι η Ευρώπη που μαθαίναμε στο σχολείο και που μας λέγανε ότι θα μπούμε στην Ευρώπη. Και εγώ είμαι από αυτή τη γενιά του 80 που η Ευρώπη ήταν θαυμάσια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Ισπανούς uh, ε, συναδέλφους και, και τα παιδιά που είναι πίσω από εμά και παρακολουθούν. Και θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, μια και μιλάμε για την Ελλάδα και την Ισπανία, ότι αυτό το μπλόκους που έχει σήμερα η Ελλάδα θυμίζει τον μπλόκο που είχε η Ισπανική Δημοκρατία ε, το 1936 και μετά. Gracias. Bueno, yo creo... Ευχαριστούμε. Αυτό που δείχνουμε εδώ είναι ότι η αριστερά θέλει τη δημοκρατία, δεν τη φοβάται. Ότι όταν η κυβέρνηση ε, ρωτάει τη γνώμη του το λέω είναι καλό. Και ότι η αριστερά δεν υποκύπτει σε ουλτιμάτουμ, σε τελεσίγραφα και σε εκβιασμούς. Είναι ένα καλό παράδειγμα για να δούμε τι μπορεί να κάνει και η αριστερά στην Ισπανία. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλαμε να σας μεταφέρουμε. Έληξε ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ναι.